Chers collègues, si vous voulez bien prendre place, nous allons pouvoir euh, ouvrir cette. Euh, Καλησπέρα σα. Qui... Θα ήθελα παρακαλώ να αρχίσουμε την έκτακτη μα αυτή συνεδρίαση. Έκτακτη μεν, φορτωμένη ημερήσια διάταξη δε. Έχετε λάβει το σχέδιο τη ημερήσια διάταξης. Ουδέν σχόλιο δεν υπάρχει, γι' αυτό και σας προτείνω να την εγκρίνουμε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 Euh, pour que nous puissions le voter lors d'une réunion extraordinaire de la commission emploi le 19 novembre à Strasbourg euh, afin de permettre θα ψηφίσουμε λοιπόν στις 19, Στρασβούργο, στις 19 ε, Νοεμβρίου στο Στρασβούργο την έκθεση του κυρίου Σέρκας με σύμφωνη γνώμη του συγητού και του σχεδόν εισηγητών. Σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό εξάμεινο, αποφασίσαμε στη τελευταία συνεδρίαση ότι θα διοργανώσουμε του χρόνου και στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης για την ανάπτυξη όχι απλές διακοινοβουλευτικές συναντήσεις, αλλά μια ολόκληρη Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα 28 με 30 Ιανουαρίου. La Commission Emploi sera... Η Επιτροπή Απασχόλησης ε, θα συμμετέχει σε αυτήν την οργάνωση και θα οργανώσει μια ημερίδα για την απασχόληση των νέων και τον κοινωνικό αντίκτυπο των προγραμμάτων προσαρμογής στις χώρες με οικονομικές δυσκολίες. Και τρίτη ανακοίνωση της Πρόεδρου, υπάρχει απευθείας αναμετάδοση της ε, συνεδρίασής μας ε, στο διαδικτύο. Περνάμε στο σημείο 3 τώρα, έκθεση Μίλαν Κάμπρνο, θα δώσω το λόγο στον συντάκτη της γνωμοδότησης για να μας ενημερώσει για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη καινοτομία με θέμα την ενεργό και υγιή γύραση. Ένα θέμα που μας αφορά όλους. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σπανίως μεν, αλλά αυτή τη φορά ε, συμφωνώ ότι η γύραση είναι κάτι που αφορά όλη την κοινωνία και όχι μόνο εμάς και σίγουρα στο μέλλον η γύραση του πληθυσμού θα αποτελέσει αποφασιστικό ζήτημα και θα επηρεάσει την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών χωρών. Έχω συντάξει γνωμοδότηση για το θέμα της ενεργούς και υγιής γύρασης. Ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Είχαμε και την έκθεση του Μάρτιν Κάσλερ για το Ευρωπαϊκό Έτος Υγιούς Γύρασης το 2012. Η γνωμοδότησή μου λοιπόν συμπληρώνει την περσινή μας προσπάθεια και φυσικά ε, συνδυάζεται και με την έκθεση της κυρίας Ομερόιτεν για τα συνταξιοδοτικά συστήματα. Σας ε, έχει μοιραστεί φαντάζομαι το σχέδιο γνωμοδότησης. Προτείνω να βρεθεί σωστή ισορροπία μεταξύ της ευρωπαϊκής προσέγγισης αφενός και της εφαρμογής αρχής της επικουρικότητας αφετέρου. Βέβαια, το θέμα αυτό θα πρέπει να το δούμε σε διάφορα επίπεδα, όχι μόνο σε εθνικό και ευρωπαϊκό, αλλά και σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, δημοτικό, αλλά και σε επίπεδο ατομικό. Γιατί την ευθύνη θα πρέπει να την αναλάβουμε όλοι. η γύραση, το γύρας δεν είναι ασθένεια. Είναι η αναπόφευκτη μοίρα όλων μας. Ούτε μπορούμε να ασφαλιστούμε κατά του γύρατος. Η γύραση είναι μια φυσιολογική διαδικασία και μια λογική συνέπεια της ανθρώπινης ζωής, μια λογική και φυσιολογική μάλλον φάση. Όλοι λοιπόν θα πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτή την αυτό το στάδιο της ζωής μας, του γύρατος. Φυσικά παραλαμβάνω την ευθύνη την αναλάβουμε όλοι για τους ηλικιωμένου, όχι μόνο οι δήμοι, οι περιφέρειες, αλλά και οι οικογένειες. Δεν μπορεί το κράτος να υποκαταστήσει την οικογένεια, θα πρέπει λοιπόν ο καθένας στο δικό του επίπεδο να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν μπορούμε απλώ να απαιτούμε εθνικά ή υπερεθνικά συστήματα να φροντίζουν, να μεριμνούν ε, για τους δικούς μας γονείς ή τους δικούς μας ηλικιωμένους. Περιμένω τις τροπολογίες σας ε, αγαπητοί συνάδελφοι και προσβλέπω σε αγαστή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ποιος θα ήθελε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διάβασα το σχέδιο γνωμοδότησης με ιδιαίτερη προσοχή. Το θέμα της ενεργούς γύρασης είναι κατά τη γνώμη μου ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Πίσω όμως από τον τίτλο του μπορεί να περιλαμβάνει πολλές ε, ιδέες ε, ή πολλές απόψεις για το τι εστί ενεργός γύραση. Σίγουρα όλοι συμφωνούμε και δεν μπορεί κανείς να διαφωνεί με την ανάγκη προάσπισης της ενεργούς της ανάγκη κοινωνικής ένταξης των πιο ηλικιωμένων. Θέλουμε οι ηλικιωμένοι να μπορούν να ε, διατηρούν τις δραστηριότητες τους καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, να ασχολούνται με θέματα που τους ε, διασκεδάζουν, που τους ικανοποιούν. Και φυσικά το δικαίωμα στην υγεία και στις υπηρεσίες υγείας και η πρόσβαση στην ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη είναι απαραίτητη για μια υγιή γύραση και μια ενεργό γύραση. Σε όλα αυτά συμφωνούμε. Και βέβαια δεν θα δεχτούμε καμία πρόταση αν αυτή της Επιτροπής που ξεκινά από την ιδέα της ενεργούς γύρες, αλλά τη χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για να παρατείνει το όριο συνταξιοδότησης. Γιατί προσπαθεί ε, να καλύψει αυτό, το, αυτό το, το στόχο της παράτασης του ορίου συνταξιοδότησης με ωραία λόγια και φημισμούς, όπως είναι αυτός της ενεργούς γύρανσης. Σίγουρα ε, το ότι είχα, έχουμε συνταξιοδότηση αυτό είναι ένα κοινωνικό κεκτημένο και η κοινωνική συμφωνία οδήγησε στην ε, εποχή που ο εργαζόμενος ε, εργαζόταν και μετά είχε, θα απολάμβανε μια εποχή που η κοινωνία θα φρόντιζε για αυτόν, η εποχή της συνταξιοδότησης τη συνταξιοδότηση μπορεί να την αφιερώσει ο καθένα για να, κάνει, να ασχοληθεί με ό,τι δραστηριότητα τον ικανοποιεί. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε στην παράταση του ορίου τη γιατί αυτό είναι σαν να στερούμε ένα θεμελιώδη δικαίωμα και κεκτημένο των εργαζομένων. Το θέμα της, ε, του δικαιώματος στη σύνταξη δεν θα πρέπει να συνδέεται με την ε, ανεργία. Γιατί στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πάρα πολλούς ε, εργαζόμενους που, πολλούς εργαζόμενους που χάνουν τη δουλειά τους, έχουμε πολλούς νέους που δεν μπορούν να βρουν δουλειά, οπότε δεν έχει νόημα να παρατείνουμε το, το όριο συνταξιοδότησης. Έτσι θα απελευθερώσουμε θέσεις εργασίας και θα επιτρέψουμε σε νέους ή λιγότερο νέους ανέργους ε, να βρουν και αυτή μια θέση απασχόληση. Αυτό και σχετικέ τροπολογίες θα καταθέσω και για την γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Ο κύριο Έρκας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω στον κύριο Κάμπρνοχ ότι μελέτησα με προσοχή το κείμενό του, βρήκα αρκετά θετικά σημεία και θα τα υποστηρίξω ανεπιφύλακτα. Για παράδειγμα, το θέμα της επένδυσης ε, στην επιμόρφωση στην... και στην κατάρτιση και των ηλικιωμένων, ε, στην εξφάλιση της πρόσβασης τους στις νέες τεχνολογίες. Καλά όλα αυτά, αλλά υπάρχει και ένα θέμα κύριε Κάμπρνοχ, που και ως προς τον τύπο και ως προς την ουσία είναι κάπως περίπλοκο. Για παράδειγμα, το θέμα της μεταρρύθμισης ε, του συνταξιοδοτικού συστήματος. Έχουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας και μάλιστα ε, ενός μέλους του ΕΛΚ, της κυρίας Όμεν Ρόιτεν. Οπότε η, η συμπερίληψη σύντομων παραγράφων, όπως η παραγράφος 6, που μιλάει για, το, για την πραγματική ηλικία σύνταξη κτλ. Πιστεύω ότι θα μας οδηγήσει σε μη καρποφόρες συζητήσεις ε, και περιτές. Άλλωστε δεν εμπίπτουν ε, στο πεδίο μια τέτοια γνωμοδότηση Προτιμώ η γνωμοδότηση αυτή να περιοριστεί στο θέμα της ενεργούς και να αφήσει τέτοια σχόλια για την ε, άλλη έκθεση που είναι η κατεξοχή έκθεση για τις ε, συντάξεις και τις μεταρρυθμίσεις συντοξιοδοτικά. Θα υποβάλουμε λοιπόν κύριε Κάμπρνοχα τροπολογίες για να εξορροπήσουμε τη γνωμοδότηση. Γιατί καλό το θέμα τη ευελιξία και τη ελαστικότητα στην αγορά εργασία, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ και τη ασφάλεια στην αγορά εργασία, Όχι ευελιξία χωρί ασφάλεια. Γιατί σίγουρα υπάρχουν δύο όψει στην μεταρρυθμίση. Δεν μα ενδιαφέρει μόνο η ευελιξία, αλλά μα ενδιαφέρει και η ασφάλεια στην αγορά εργασία. Σε ό,τι αφορά τι νέε μορφέ εργασία δεν μπορούμε απλώς να τις ε, καταπίνουμε χωρίς κανένα σχόλιο. Θα πρέπει να τις ε, συνοδεύσουμε με διάφορα άλλα μέτρα, γιατί ένα θέμα τέτοιο είναι ευαίσθητο και για τους εργοδότες και για τους εργαζόμενους. Ανάμεικτα λοιπόν συναισθήματα για την γνωμοδότηση του κυρίου Κάμπνοχ. Με μερικά σημεία συμφωνούμε, όπως είπα, αλλά και για μερικά θα καταθέσουμε τροπολογίες γιατί δεν μας βρίσκουν σύμφωνος. Πάντως όλα αυτά θα γίνουμε πολύ επικοδομητικό πνεύμα. Ευχαριστώ. Εσύ. Θα σε ευχαριστώ. Αν δεν ζητά κάποιος άλλος το λόγο, θα ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή. Θα σε ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δύο λόγια μόνο. Συμπερασματικά, όσον αφορά τον αριθμό των παρόντων, διαπιστώνω ότι ίσως ε, το θέμα της γύρανσης με ενεργό και υγιή τρόπο δεν είναι κάτι που θεωρείται προτεραιότητα εδώ. Άκουσα πολύ προσεκτικά αυτό που είπατε όσον αφορά την δυνατότητα συμμετοχής σε εργασίες, πρόσβαση στον αθλητισμό, σε πολιτιστικές δραστηριότητες, καθώς και τον σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει η πρόβλεψη, η πρόγνωση κυρίως ε, στον τομέα της υγείας. Καθότι ενεργός γύρανση και υγιής γύρανση σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να ζήσει ανεξάρτητα και να υποφεληθεί από όλες τις ε, κοινωνικές υπηρεσίες που προσφέρει. Βεβαίως, Με μεγάλη χαρά θα εξετάσω τροπολογίες που αφορούν την ελαστικότητα αλλά και την ασφάλεια της αγοράς εργασίας. Αλλά σαφώς θα πρέπει να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων και των εργοδοτών. Ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Προθεσμία 12 Μαΐου. Όχι, Νοεμβρίου λέει ο Πρόεδρος στις 12. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες στις 28 και 29 Νοεμβρίου. Στα αγγλικά πρέπει να υποβληθούν οι τροπολογίες. Και από τις 12 ως 28 Νοεμβρίου θα μεταφραστούν. 28-29 Νοεμβρίου εξετάζονται λοιπόν οι τροπολογίες συμβιβαστικές στις 6 Δεκεμβρίου και ψηφίζουμε αμέσως μετά. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ψηφίζει στις 18 Δεκεμβρίου. Σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Η συγγήτρια δεν είναι παρούσα. Τι να σας πω. Και εμείς έχουμε ψηφοφορίες. Ας προχωρήσουμε λοιπόν με τα δύο επόμενα σημεία, αφού δεν είναι παρούσα το σημείο 5, Γιούτε Steinrück, η οποία θα μας παρουσιάσει το θέμα των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο σχετικά με το πρόγραμμα με το Συμβούλιο, ε, με το Συμβούλιο, συγγνώμη, σχετικά με το πρόγραμμα για την κοινωνική αλληλεγγύη και καινοτομία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ναι, έγινε ο πρώτος γύρος των ε, διαπραγματεύσεων, ο οποίος ε, και όσον αφορά τη δική μου άποψη, αλλά και από όσο άκουσα από τους και ηγητές, ήταν απογοητευτικός. Δεν ελήφθησαν καθόλου σοβαρά υπόψη τα κεντρικά σημεία που είχε υποβάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον αφορά την μικροχρηματοδότηση, ξεκίνησε η συζήτηση προς κάποια κατεύθυνση, μπορούμε να πούμε ικανοποιητικά, Αύριο θα υπάρξει η δεύτερη συνάντηση, τριμερής. Θα ξεκινήσει κατά την άποψή μας εκεί η πραγματική διαπραγμάτευση και θα ακολουθήσει μια ε, δήλωση. Η πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την ε, μεταρρύθμιση ε, όρους κατά την άποψή μας ε, θα πρέπει να ξανασυζητηθεί και περιμένουμε να αποσαφηνίσει η Επιτροπή κάποια από τα σημεία. Επαναλαμβάνω, ε, η εργασία των σκιωδών εισηγητών ήταν εξαιρετική και όλα έγιναν σε ένα πνεύμα πολύ καλής συνεργασίας. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο για το θέμα αυτό. Εγώ ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια γιατί πρόκειται για μια δύσκολη διαπραγμάτευση και το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ μας είναι καθοριστικό σε μια τέτοια διαπραγμάτευση. Εμείς έχουμε καθορίσει και θέσει τις προτεραιότητές μας, ιδιαίτερα για θέματα όπως η μικροχρηματοδότηση που έχει προτείνει το Συμβούλιο. Τελικά, πιστεύω θα αντιμετωπίσουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στη συζήτηση για τους νέους. Εμείς θελήσαμε να το θέσουμε σαν προτεραιότητα σαν προϋπόθεση. Από ό,τι είδαμε όμως το Συμβούλιο απάντησε ότι αρνείται να συζητήσει το θέμα αυτό σε αυτή τη βάση και εμείς αναγκαστήκαμε εδώ να τηρήσουμε μια σκληρή στάση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την εισηγήτρια γιατί μπορέσαμε να κάνουμε ικανοποιητικά βήματα. Η κυρία Μακίνητη δεν είναι εδώ, δεν γύρισε ακόμα, ούτε η κυρία Μογάν Σαχτιέ. Είμαι λοιπόν σε δύσκολη κατάσταση. Δυστυχώς, και δεν με ευχαριστεί αυτό, θα αναγκαστούμε να διακόψουμε ως τις 4 και 4. Και ζητώ συγγνώμη προς όλους όσους ήρθαν στην αίθουσα, περίμεναν να συζητήσουν την έκθεση της κυρίας Μαρκίντερ. Ζητώ συγγνώμη επίση και τους διερμηνείς και ελπίζω ότι θα τελειώσουμε στην ώρα μας παρόλη την καθυστέρηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας προτείνω να συνεχίσουμε. Έχει έρθει στο μεταξύ κυρία Μακιντάιρ. Οπότε ας περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης παρακαλώ και να δώσουμε το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Μακιντάιρ, για να μας παρουσιάσει τις 44 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για το σχέδιο γνωμοδότησής της που ε, θα υποβληθεί στην ε, Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και έχει θέμα τη βελτίωση τη πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ που αναβάλατε τη συνεδρίαση και μου επιτρέψατε να ψηφίσω στην Επιτροπή Ελευθεριών πριν έρθω εδώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους κατέθεσαν τροπολογίες για την γνωμοδότηση αυτή. Έχουμε 44 τροπολογίες και ομολογώ ότι υποστηρίζω τις περισσότερες. Υπάρχουν κάποιες που δεν μπορώ να στηρίξω και υπάρχουν και κάποιες πάνω στις οποίες χρειάζομαι κάποιες διευκρινήσεις. Εκτιμώ το ότι έχουν φέρει φρέσκες ιδέες και ελπίζω ότι θα συμβάλλουν στο να γίνει μια καλή γνωμοδότηση. Θα προτείνω και κάποιες συμβιβαστικέ ε, τροπολογίες και θα τις κυκλοφορήσω πριν από τη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών αύριο Μόνο δύο-τρία σημεία θέλω να θίξω. Καταρχήν, έχει μεγάλη σημασία να μην επαναλάβουμε τις εργασίες της Επιτροπής Ελευθεριών. Υπάρχουν πολλοί τομείς που μπορούμε να συζητήσουμε τα θέματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά πρέπει πάνω απ' όλα να συζητήσουμε τις δικές μας. Small businesses, micro businesses particularly hard. Ε, με συγχωρείτε, δεν, Lead Committee, όχι η Επιτροπή Ελευθεριών. Πολλές από τις εταιρείες υποφέρουν από την οικονομική δυσχέρεια και ξέρουμε πως χάνονται πολλές θέσεις εργασίες. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες επιλογές έχουμε. Ε, πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση των τραπεζών. Ε, χρειαζόμαστε, υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες στον Ευρωπαϊκό Ορίζοντα, το Horizon και άλλα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε για να ενισχύσουμε τις δυνατότητες και να ενισχύσουμε και τους επιχειρηματίες με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την υγιή οικονομική διαχείριση των εταιριών τους, των επιχειρήσεών τους, έτσι ώστε να έχουν την τεχνογνωσία να βρίσκουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Γιατί μόνο βρίσκοντας πρόσβαση στη χρηματοδότηση μπορούν να αυξηθούν, να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν καινούριε θέσεις εργασίας. Ε, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μου και αναμένω να συνεργαστώ και με τους σκιώδεις συζητητές αύριο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ την εισηγήτρια για την, το πολύ καλό κείμενο βάσης που μας έχει δώσει. Ε, συμφωνώ με αυτά που είπε ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βρίσκουν χρηματοδότηση γρήγορα και άμεσα από τις τράπεζες. Και εδώ ε, ειδικά τον καιρό της κρίσης και ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό που μερικές φορές είναι ο κανόνας για τις τράπεζες. Δηλαδή η τράπεζα αυτό που λένε ότι σου δίνει μία ομπρέλα όταν δεν βρέχει και όταν βρέχει σου λέει συγγνώμη δεν έχω μπρέλα να σου δώσω πρέπει να βραχείς. Αυτό δεν πρέπει να γίνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, τώρα εγώ προέρχομαι και από την Ελλάδα. Ξέρετε όλοι ε, πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Ξέρετε όλοι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και αντιλαμβάνεστε όλοι πόσο μεγάλη ανάγκη έχουν από χρηματοδότηση και οι ελληνικές αλλά όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στην Ευρώπη. Ε, με αυτή την έννοια ε, συμφωνώ με την εισηγήτρια και το γενικό της πνεύμα. Προσπάθησα και εγώ να είμαι δημιουργική και έχω καταθέσει αρκετές τροπολογίες. δεν θα επεκταθώ εδώ για να αναλύσω τις τροπολογίες, μη σας κουράσω, να είμαι σύντομη. Ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία, αυτό μόνο θα πω, η ενημέρωση. Να ξέρει ο ιδιοκτήτης της μικρομεσαίας επιχείρησης πού μπορεί να απευθυνθεί για να πάρει πληροφορίες, να ξέρει τους μηχανισμούς τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιήσει για να βρει κεφάλαια. Ε, περιμένω με ανυπομονησία τις συμβιβαστικές και θα είμαι αύριο στη συνάντηση βεβαίως που θα κάνουμε η για να δουλέψουμε όσο καλύτερα γίνεται και πιο αποτελεσματικά για τους Ευρωπαίους πολίτες που έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και που θέλουμε να τις στηρίξουμε. Ευχαριστώ. Merci, euh, Nadia Hirsch. Thank you, Madam Chair. Uh, on behalf Θα ήθελα εκ μέρου του σκιώδου συγκεκριτού μα ε, να υποβάλω κάποιε παρατηρήσει. Να ευχαριστήσουμε καταρχήν ε, την εισηγήτρια για το έργο τη. Είναι ένα έγγραφο που επισημαίνει τα βασικά προβλήματα που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση. Και σίγουρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι οι μεγαλύτεροι εργοδότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό θα πρέπει να τις υποστηρίξουμε, γιατί αυτές δημιουργούν πολλές θέσεις απασχόλησης. Γνωρίζουμε τι τεράστιο δυναμικό έχουν για να αντιμετωπίσουν χρόνια προβλήματα όπως είναι η ενέργεια των νέων, όπως είναι το κενό που υπάρχει στις ειδικευμένες θέσεις εργασίας και στην προσφορά ε, μαθητείας ε, ή διαφόρων μηχανισμών ε, εκμάθησης και κατάρτισης. Έχουμε διάφορες τροπολογίες από το σκιώδη συγγητή. Έχει τονιστεί ότι πολλές φορές ε, τα επιτόκια δανεισμού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αποτρεπτικά υψηλά και γι' αυτό είναι δύσκολη η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Επίσης ε, και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα μπορούσαν να, ε, να θεσπίσουν τις δικές τους επενδυτικές τράπεζες και να προωθήσουν την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και γενικώ του κλάδου των μικρών επιχειρήσεων. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάτι κάτι σαν αυτό που υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο πράσινες επενδύσεις, να στηρίξουμε συνεταιρισμούς ή άλλους τομείς που αποκλείονται από τις ε, κεφαλαίκες επενδύσεις. Ο σκιώδης ηγετής μας προσβλέπει σε συνεργασία με τους συναδέλφους και φαίνεται από τις διάφορες τροπολογίες ότι υπάρχει δυναμικό και βάση για καλές συμβαστικές τροπολογίες στα περισσότερα από τα κέρια ζητήματα της γνωμοδότησης κυρία Ζουμπέρ θα ήθελα να πω ότι υπάρχει γενική σύμπνοια και συμφωνία για τη γνωμοδότηση και εμείς καταθέσαμε κάποιες τροπολογίες. Ε, μερικές είναι πιο λεπτομεριακές, άλλες είναι πιο γενικές. Θα πρέπει σίγουρα να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις πολύ μικρές επιχειρήσεις ε, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα COSME προτείνουμε και οι μεσαίες επιχειρήσεις ε, να ε, εποφεληθούν από την αύξηση της, από την ενίσχυση της πρόσβασης ε, στη χρηματοδότηση και πιστεύω ότι η πρόσβαση χρηματοδότηση για τους συνεταιρισμούς και για τις κοινωνικές επιχειρήσεις θα να, τη χάνει κάποια ρύθμισης γιατί εμπίπτει σε διαφορετικό πλαίσιο από αυτό που ισχύει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ήθελα όμως εδώ να επισημάνω και μερικά ουσιαστικά θέματα. Είναι προφανές ότι ε, συμφωνούμε πως η τράπεζα υποχρεούται να χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονομία. Αυτό, αυτό το σκοπό θα πρέπει να υπηρετούν οι τράπεζες, να εξυπηρετούν την κοινωνία, την πραγματική οικονομία. Και σίγουρα οι τράπεζες ε, έχουν λάβει έναν πακτολό κρατικό κονδύλιο και μάλιστα πολλά από αυτά πήγαν χαμένα. Όσοι γνωρίζουν τον κόσμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, γνωρίζουν ότι το βασικό τους πρόβλημα προέρχεται από, την, ε, από τις χαμηλές κρατικές επενδύσεις και τον περιορισμό της ιδιωτικής κατανάλωσης. Οπότε, αν δεν ε, θεσπιστούν κάποια μέτρα για την τόνωση της κατανάλωσης, δεν πρόκειται να βοηθηθούν οι, μικρομεσαίες, επιχειρήσεις ώστε να εξασφαλίσουν μια βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους. Η Πρόεδρος. Ωραία. Δεν θέλει άλλο κανεί το λόγο. Δεν ξέρω αν η συγκεκριά μας η κυρία Μακιντάιρ θέλει να δευτερολογήσει. Την επόμενη φορά θα μας καταθέσετε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες και σας ευχόμαστε καλές διαπραγματεύσεις. Το σημείο 5 το α, διεκπαιρεώσαμε. Για το σημείο 6 η κυρία Μωράν είναι απουσιάζει. Μου ανέθεσε ε, την ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Να σας πω ότι στις 5 Ιουλίου ψηφίσαμε για την διαπραγματευτική εντολή. Στις 19 Ιουλίου έγιναν προπαρασκευαστικές ε, συνεδριάσεις και μέχρι στιγμής είχαμε τρεις ε, τριμερεί διαλόγου, 18 ε, Σεπτεμβρίου και 2 τον Οκτώβριο. Συμφωνήσαμε να περιοριστούμε σε θεματολογικές, θεματικές ενότητες. Αυτό ζήτησε και το Συμβούλιο για να οργανώσουμε εκ τη συζήτηση για τον ειδικό κανονισμό για το κοινωνικό ταμείο και τον οριζόντιο κανονισμό για το οποίο είναι κατ' ουσία αναρμόδια η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Και με βάση την ενισχυμένη συνεργασία για το θέμα αυτό, η συγκεκριτής μας είναι ο κύριος Κοζά. Σε ό,τι αφορά την ε, διαπραγματευτική θέση του Συμβουλίου, αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη επίσημα διαπραγματευτική εντολή, κάτι που περιπλέκει κάπως τις διαπραγματεύσεις και τις καθιστά και πιο συναρπαστικές. Οπότε το Συμβούλιο στηρίζεται σε μια γενική δική προσέγγιση. Το όνομα τα λέει από μόνο, μιλάει από μόνο του. Είχαμε τον Απρίλιο-Ιούνιο και τον Οκτώβριο τρει τρεις ε, συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Η θέση αυτή όμω δεν καλύπτει το σύνολο του κανονισμού και θα πρέπει να συμπληρωθεί ιδιαίτερα για το άρθρο 2, για τις εκπομπές και το 15 για, τα, για τους χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς ε, θα συμπληρωθεί αργότερα. Οπότε η εξέταση των ε, τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν πέρασε από διαπραγμάτευση, ούτε συζητήθηκε ε, διεξοδικά από το Συμβούλιο. Μια και η Κυπριακή Προεδρία περιμένει από το Κοινοβούλιο να εξετάσει το σύνολο και να υποβάλει μία συγκροτημένη θέση ε, για το σύνολο της πρότασης. Ενώ εμείς ε, εξετάζουμε αναενότητα τη θέση του Συμβουλίου και περιμένουμε ε, την ολοκλήρωση του πακέτου για να διαμορφώσουμε τη γνώμη μας. Η Κυπριακή Προεδρία επίσης δεν θέλει να επισημοποιήσει την πρόοδο που έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμή στις διαπραγματεύσεις με βάση την παλιά μέθοδο ότι δεν υπάρχει συμφωνία για κανένα σημείο αν δεν, αν επιτευχθεί συμφωνία για το σύνολο. Σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό είχαμε οριστικοποίηση κάποιων άρθρων υπό την επιφύλαξη βέβαια της ε, επισημοποίησης και της θέσης του Συμβουλίου και τα άρθρα για τα οποία έχουμε καταλήξει συμφωνία είναι τα άρθρα 6 για τη συμμετοχή των εταίρων, άρθρο 7 για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, το άρθρο 8 για την ισότητα ευκαιριών και τη μη διακριτική μεταχείριση, άρθρο 9 ε, κοινωνική καινοτομία, άρθρο 10 για τη διασυνοριακή συνεργασία, άρθρο 11 που περιλαμβάνει ειδική συζήτηση για τα επιχειρησιακά προγράμματα, και το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότηση μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τώρα, για ποια σημεία υπάρχουν διαφωνίες. Διαφωνίες υπάρχουν κυρίως ότι η γενική ειδική προσέγγιση του Συμβουλίου καθιστά προαιρετική για τα κράτη-μέλη, προαιρετικό για τα κράτη-μέλη ένα μεγάλο τμήμα των υποχρεώσεων που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να γίνουν ε, δεσμευτικές, όπως προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό ισχύει για, μια τροπολογία που λέει ότι μόνο 2% των ε, πόρων στις περιοχές Α και Β ε, αφιερώνεται στη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις δράσεις του ΕΚΤ ή σε βελτιώσεις της ισότητας των δύο φύλων και στην καταπολέμηση των διακριτικών μεταχειρήσεων. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν για όλα τα επιμέρους σημεία και φυσικά θα σας ενημερώνουμε στο μέτρο των εξέλιξεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, τις ε, με το Συμβούλιο, δεν υπάρχουν ε, αρκετές ημερομηνίες συνεδρίασης. Πάντως, η προκαταρκτική συμφωνία περιλαμβάνει μόνο ένα σημείο και μία τροπολογία, μία συμβαστική τροπολογία που και αυτή χρήζει διευκρινή στα πλαίσια του γενικού κανονισμού. Το δεύτερο τώρα πακέτο, για το οποίο ξεκινήσαμε τη συζήτηση, είναι αυτό που αφορά τη θεματική συγκέντρωση. Ένα ευαίσθητο σημείο στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Αφορά τα άρθρα 3 και 4 της πρότασης. Μάλιστα, μέχρι στιγμής μόνο μία τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πακέτο αυτό έχει συζητηθεί και δεν έχει ενταχθεί σε καμία συμβαστική τροπολογία. Νομίζω ότι σας παρουσίασα πιστά την ε, μέχρι τώρα κατάσταση και τις εξελίξεις από τις διαπραγματεύσεις. Όσοι συμμετέχουν σε τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις ε, ξέρουν ότι το κλειδί της επιτυχίας έγκυται στην υπομονή, στην αποφασιστικότητα και στην ε, μεθοδικότητα, αρετές που είμαι βέβαια ότι θα επιδείξει η διαπραγματευτική μας ομάδα. Αυτά τώρα και περνάμε στο σημείο 7, στις ψηφοφορίες δηλαδή. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Έπρεπε να σας είχα προτείνει συζήτηση για την ενημέρωση αυτή ως προς τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Κανένα πρόβλημα, κυρία Πρόεδρε. Απλώ ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι η Επιτροπή μας είναι κατ' ουσία αρμόδια για την έκθεση για τις χερσαίες μεταφορές. Δυστυχώς απουσίασα ε, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, γιατί είμαστε στην Επιτροπή Μεταφορών. Έχουμε πια την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σας διαβεβαίω ότι ήταν πολύ θετική έκβαση στην Επιτροπή Μεταφορών. Απλώς ήθελα να σας ενημερώσω για αυτή την τελευταία εξέλιξη. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Σιγητά. Συγγνώμη, δεν ε, φανταζόμουν ότι θα έχετε τέτοιες χαρμόσυνες ειδήσει. Ελπίζω να μην είναι και οι τελευταίες. Τώρα, περνάμε στο σημείο 7. Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης υπομορφήν επιστολής για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και ενεργοποίηση του Ταμείου αυτού για την ε, βιομηχανία κατασκευής μοτοσυκλετών στην Εμίλια Ρωμάνια της Ιταλίας. Ποιος είναι υπέρ? Κατά αποχές Εγκρίνεται λοιπόν ε, η γνωμοδότηση αυτή υπό μορφή επιστολή. Δεύτερη κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση αφορά την υπόθεση Νόκια από τη Φιλανδία. Ποιο είναι υπέρ κατά τη επιστολής, αποχέ. εγκρίνεται και αυτή η επιστολή. Σημείο 9 και πάλι τρίτη αίτηση κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμόγης στην Παγκοσμιοποίηση και πάλι για την Όκια στη Ρουμανία όμω. Θα ήθελα για να διευκρινίσω σε όσους δεν είχαν το προνόμιο να συμμετέχουν στο, στην ομάδα πρόκειται για κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ε, για μια περίπτωση που αφορούσε με την κατάσταση ενός εργοστασίου από την Γερμανία στη Ρουμανία. Ήδη είχαμε τέτοια υπόθεση στο παρελθόν, τώρα συνεχίζεται η προσπάθεια υποστήριξης των εργαζομένων της Νόκια στη Ρουμανία, γιατί το εργοστάσιο που είχε προγραμματιστεί να κατασκευαστεί στη Ρουμανία, τρία χρόνια μετά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η κατασκευή του. Γι' αυτό και υποβάλλει τη δεύτερη αίτηση για την ενεργοποίηση του Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Αυτή τη φορά η Νόκη αποφάσισε να μετεγκατασταθεί στην Ασία. Ποιο είναι υπέρ τη επιστολής. Κατά, απόχέ. εγκρίνεται και η επιστολή αυτή. Τέταρτο αίτημα ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση αφορά μια περίπτωση στην Αυστρία που σε περιφερειακό πλαίσιο ζητήθηκε η ενεργοποίηση του Ταμείου για να βοηθηθούν οι κοινωνικοί λειτουργοί μετά την θέσπιση προγράμματος λιτότητας που αποφάσισαν οι περιφερειακές αρχές της Αυστρίας. Στην περίπτωση αυτή έχουμε δύο τροπολογίες του ΕΛΚ που καλούμαστε να ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε πρώτα την πρώτη τροπολογία του ΕΛΚ που θεωρεί ουσιαστικά ότι οι απολύσεις αυτές δεν σχετίζονται με την κρίση. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η τροπολογία. Αλλά ας γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος. Καταρχήν έχετε όλες τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας. Ναι, από ό,τι φαίνεται άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 16 υπέρ, 19 κατά και 4 αποχές. Απορρίπτεται όντως η τροπολογία αυτή και περνάμε στη δεύτερη τροπολογία του ΕΛΚ ε, την υπέβαλε η κυρία Μπάουερ εκ μέρου του ΕΛΚ για την προσθήκη νέα παραγράφου, της παραγράφου 8, που λέει ότι δεδομένου του, του ποσοστού επιδοτήσεων και επιδοτήσεων κατάρτισης ε, που είναι αδικαιολόγητες. Ε, ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας αυτής κατά αποχές μάλλον εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας. 22 υπέρ 16 κατά όντως είχε εγκριθεί τροπολογία και ψηφίζουμε το σύνολο της επιστολής όπως έχει τροποποιηθεί. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, τέλος. 23 υπέρ, 13 κατά και 4 αποχές. Εγκρίνεται και η επιστολή αυτή. Ερχόμαστε τώρα στην πέμπτη περίπτωση κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου, εδώ έχουμε μια περίπτωση από τη Δανία. Θέτω σε ψηφοφορία το σχέδιο της επιστολής. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έκτη περίπτωση. Μεταλλουργία. Κινητοποίηση λοιπόν στην Ισπανία. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτή η επιστολή. Τελευταία περίπτωση πρόκειται για μια απόλυση στην εταιρεία ΣΑΜΠ. Ε, η αίτηση, το αίτημα υποβλήθηκε από την Σουηδία, Σουηδία που είναι κατά της ε, επέκτασης του κριτηρίου της κρίσης ε, και έτσι δικαιολογείται η κινητοποίηση του Ταμείου. Ποιοι είναι υπέρ. ναι, ναι, για τους εργαζόμενους, αλλά είναι η κυβέρνηση που υπέβαλε το αίτημα για την κινητοποίηση του Ταμείου. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Αυτή η έβδομη και τελευταία επιστολή, λοιπόν, εγκρίνεται. Ερχόμαστε, λοιπόν, τώρα... Το σημείο 14 και θέτω σε ψηφοφορία την έκθεση της κυρίας Μάριαν Χάρκιν για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Πρόκειται για ένα κείμενο νομοθετικού περιεχομένου με βάση το πολιετές ε, οικονομικό πλαίσιο. ...299 τροπολογίες πρόκειται να εξετάσουμε έξι γνωμοδοτήσεις, γνωμοδότηση και της Επιτροπής για τα Γεωργίας με βάση το άρθρο 4.3 στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας. Η Ωστόσο απορρίφθηκε αυτό το κείμενο, δεν μπορούμε να το εξετάσουμε και υπάρχει μια συμβιβαστική... θα πρέπει να έχουμε συμβιβαστική τροπολογία. Έχει υποβληθεί μία από τους και θα πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, πριν από το σημείο 1... Je vais mettre voix l'amendement 54. Θέτω σε ψηφοφορία την τροπολογία 54 που είναι μια πρόταση απόρριψης. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, δεν εγκρίνεται. Σε ψηφοφορία την 226. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρθρο 1. Μετά την παράγραφο 1. Συμβιβαστική ΑΕΦ από πέντε ομάδες, 5 πολιτικές ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 1, παράγραφος 2. Ε, ε, πάλι οι πέντε ίδιες πολιτικές ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε unblock ε, το 1, που είναι η συμβιβαστική τροπολογία 1H και 1G. Πέντε πολιτικές ομάδες από πίσω. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνούμε λοιπόν στο άρθρο 1 μετά την υποπαράγραφο 2, θέτουμε σε ψηφοφορία την παράγραφο 8 από την ε, Επιτροπή Ίντα Εσωτερικών Υποθέσεων. Υπέρ, κατά, αποχές. Θέλετε να ξαναρχίσουμε. Ποιοι είναι υπέρ για την 8 από τις Επιτροπές Εσωτερικών Υποθέσεων. Κατά, αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 1, παράγραφος 3. Συμβιβαστική τροπολογία L. Από πολύ περισσότερες πολιτικές ομάδες. 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 3 μετά το πρώτο εδάφιο, καινούριο σημείο, συμβιβαστική τροπολογία ΑΕ, από πέντε πολιτικές ομάδες. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο Α, αίμα, τέσσερις πολιτικές ομάδες. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο Β, ε, συμβιβαστική πρόταση 1, νη, τέσσερις πολιτικές ομάδες, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο Γ. Θέτουμε σε ψηφοφορία πέντε ταυτόσιμες ε, τροπολογίες, τη 16 της εισηγήτριας, την 144 της κυρίας Ζούμπερ, την 145 της κυρίας Κορνέλισεν, την 146 της κυρίας Ούμεν Ρούιτεν, την 147 του κυρίου Μπουλάν. Πέντε λοιπόν για κατάργηση κειμένου. Υπέρ, κατά, αποχές, υπερψηφίζονται αυτές οι πέντε τροπολογίες κατάργησης κειμένου. Θέτουμε σε ψηφοφορία... Ένα. Alors, l'amendement 1 est couvert et donc nous n'avons pas besoin de le voter. Δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε μάλλον αυτή. Οπότε, α όχι, πρέπει να το ψηφίσουμε το μπλοκ 2. Όχι, όχι, δεν μπορεί να ψηφιστεί. Pardon.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 Ζητώ συγγνώμη. Η συμβιβαστική πρόταση AM εισαγάγει ένα καινούριο σημείο, άρα δεν μπορεί να καταργηθεί φυσικά. Επομένως, τη θέτω σε ψηφοφορία. Υπέρ της AN. Υπέρ. Κάτα. Άποχες. Φοβάμαι ότι έχει απορριφθεί, αλλά θα επαληθεύσουμε αν το ζητήσει ο κύριος Νταρντά. Ναι, θα επαληθεύσουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 13 υπέρ, 22 κατά, 5 αποχές. Επομένως, αυτή η συμβιβαστική τροπολογία απορρίφθηκε. Ερχόμαστε τώρα στο μπλοκ υπαριθμών 2. Υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται το μπλοκ 2. Θέτω σε ψηφοφορία το μπλοκ 3. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 3. Καλύφθηκε από το μπλοκ, επομένως ερχόμαστε στο άρθρο 4, παράγραφος 1α, τροπολογία 163 της κυρίας Μπιζότο. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές, απορρίπτεται. 164 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 165 της κυρίας Μπλίνκεβιτσι Τζιούτε. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άρθρο 4, παράγραφος 1β. Θέτουμε σε ψηφοφορία την τροπολογία 167 της κυρίας Μπιτζότο. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 17 της Επιτροπής Περιφερειών. Υπέρ, κατά, αποχές νομίζω πως έχει απορριφθεί, αλλά θα κάνουμε έλεγχο. 17 της Επιτροπής Περιφερειακών Υποθέσεων. Ψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 17 υπέρ, 24 κατά. Δεν εγκρίνεται. Επομένως, θέτουμε σε ψηφοφορία την 168. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 166 τη κυρία Κορνέλισεν υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο βα, καινούριο, τροπολογία 170, ζουμπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Άρθρο 4, παράγραφος 2. Πρόκειται για δύο ταυτόσιμες προτάσεις, η παράγραφος 3 της Επιτροπής ε, Εσωτερικών Υποθέσεων και 18 της Επιτροπής Περιφερειακών Υποθέσεων. Τις θέτω σε ψηφοφορία μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 4, παράγραφος 3. Καλύφθηκε αυτό. Επομένως, τώρα θέτουμε σε ψηφοφορία το άρθρο 5, παράγραφος 1α, τροπολογία 21 της εισηγήτριας και 182 Σούμπερ που είναι ταυτόσιμες. Article 6, Με συγχωρείτε, άρθρο 6, παράγραφος 1α, τροπολογία 21 και 192, διορθώνει η πρόεδρος δύο ταυτόσιμες τροπολογίες. Τις θέτουμε σε ψηφοφορία από κοινού. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 7, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1, εισαγωγικό τμήμα, 198 σούπερ, 199 μπενιών, τις θέτουμε σε ψηφοφορία μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συνεπία αυτού ε, καταπίπτει η τροπολογία 16, οπότε θέτω σε ψηφοφορία το άρθρο 6, παράγραφος 1, γάμα, παράγραφος 15 της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ, υπέρ. Κανονικά η εισηγήτρια είναι κατά. 15 είναι άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο εδάφιο γάμα. καταπίπτει η 16 της ίντα. Βρισκόμαστε στην 15 της ίντα. Σας βεβαιώνω ότι εκεί βρισκόμαστε. 15. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, δεν εγκρίνεται. Άρθρο 7, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1, εδάφιο α, συμβιβαστική τροπολογία R, με από πέντε πολιτικές ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 7, παράγραφος 1, υπό παράγραφος 1, εδάφιο Β, ε, συμβιβαστική τροπολογία S από τέσσερις πολιτικές ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 7, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1, εδάφιο γ, εισαγωγή του σημείου, παράγραφος 10 της Επιτροπής Γυναικών, υπέρ. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρθρο 7, παράγραφος 1, καινούρια παράγραφος, από τέσσερις ε, πολιτικές ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται η AG. Άρθρο 7, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2, συμβιβαστική τροπολογία AM από τέσσερις πολιτικές ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 7, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 3, συμβιβαστική λύση T από τέσσερις πολιτικές ομάδες υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 7, παράγραφος 2, σημείο α, τροπολογία 218 της κυρίας Edith Bauer, υπέρ, καλτά, αποχές, νομίζω πως έχει εγκριθεί, αλλά θα κάνουμε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. 2.18 της κυρίας Bauer, πέρας της ψηφοφορίας, 24 υπέρ, 17 κατά, εγκρίνεται. Άρθρο 7, παράγραφος 2, μετά από το σημείο α, συμβιβαστική λύση AK από 4 πολιτικές, 5 πολιτικές ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 7, παράγραφος 2, σημείο Β, τροπολογία 219 της κυρίας Κορνέλησεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 της συγκέντριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 7, παράγραφος 3, Συμβιβαστική λύση U από πέντε πολιτικές ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 παράγραφος 1 από τέσσερις πολιτικές ομάδες. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 8. Παράγραφος 2, 2, 1. W, συμβιβαστική. Πέντε ομάδες. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8, 8 παράγραφος 2, εδάφιο 1, νέο, με μια τροπολογία 230 της κυρίας εν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρθρο 8, παράγραφος 2, εδάφιο α. Πρόκειται για την 27 τροπολογία της Επιτροπής Περιφερειών. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 8, παράγραφος 2, νέο β. Πρόκειται την τροπολογία 231 της κυρίας Μπιζότο, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8, άρθρο 8, παράγραφος 2, γάμα, σι, πρόκειται για την 232, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8, 2, ε, πρόκειται για 31, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται και μετά το ε πρόκειται για την τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 8 παράγραφος 2G πρόκειται για την συμβαστική Χ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και μετά το G παράγραφος 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και στο H, συμβαστική Y υπέρ κατά αποχές υιοθετείται αυτή η συμβαστική τροπολογία. Στο σημείο I, 35 υπέρ κατά. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 35 κατά αποχές εγκρίνεται. 235 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 8 παράγραφος 2 παράγραφος I νέο πρόκειται για τη συμβαστική α λάμδα AL ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Άρθρο 8 παράγραφος 3 νέα τροπολογία 238 της κυρίας Μπλίνκεβιτς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9, παράγραφος 1. Τροπολογία 37 τη ηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 9, παράγραφος 2. 37 Επιτροπής Πληροπολογισμών υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε. Τέλος. 25 υπέρ, 16 κατά. Εγκρίνεται η 37. Παράγραφος 32 της περιφερειακής υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 παράγραφος 3. Πρόκειται για την 239 της κυρίας Κονέλσεν υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 9 παράγραφος 4. Είναι η παράγραφος 38 της Επιτροπής Προπολογισμών υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 9, μετά την παράγραφο 4, τροπολογία 240 Κονέλησεν, υπέρ. Θέλετε να επαληθεύσουμε το 38 της Επιτροπής Προπολογισμών. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε την 38. Ψηφίσατε όλοι, τέλος. 29 υπέρ, 9 κατά. Και τρεις αποχές. Κάτι έγινε εδώ. Ήταν απαραίτητο λοιπόν να επαληθεύσουμε. 240 τροπολογία της κυρίας Κονέλης είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα ελέγξουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. 16 υπέρ, 24 κατά. Κυρία Κονέλησεν, λυπούμε, αλλά απορρίφθηκε η τροπολογία σας. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 9, συμβαστική Ζ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνει. Και τώρα πάμε στο άρθρο 10, συμβαστική ΑΑ, 6 ομάδες την υποστηρίζουν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 11, πράγματος 1, 241, τροπολογία Κορνέλησεν. Θα ψηφίσουμε σε δύο τμήματα. Το σύνολο του κειμένου χωρίς την λέξη ΕΣΑΦ. Υπέρ, κατά, αποχές, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Το πρώτο τμήμα. 17 υπέρ 23 κατά απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα δεν έχει πλέον νόημα. Άρθρο 11 παράγραφος 4 συμβαστική αλφαβήτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 12 τίτλο πρόκειται για την 245 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 12 παράγραφος 1 η 246 Κορνέλησεν υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άρθρο 12, παράγραφος 2, 40 της κυρίας Αρκίν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 12, παράγραφος 3, συμβιβαστική AC, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 12, παράγραφος 4, τροπολογία για εξάλληψη της κυρίας Μπιζότο, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 250, Κορνέλισεν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 13, παράγραφος 1. Ψηφίζουμε. Το μπλοκ 4, συμβιβαστική α, δ και η. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα φτάνω στο άρθρο 13, παράγραφος 1, σημείο Δέλτα, νέο, τροπολογία 230, συγγνώμη, 266, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άρθρο 13, παράγραφος 3, 37 της περιφερειακής υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε την 267 τροπολογία υπέρ. Υπέρ κατά αποχές. Άρθρο 14. Συγγνώμη, 268. Η 44 έχει ψηφιστεί. Και πάμε στην 15, άρθρο 15, παράγραφος 2, παράγραφος 2, νέο, παράγραφος 24 της ίντα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 15, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 1, 45 της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Υπέρ εισηγήτρια. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 15, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 2, 46 της ε, Επιτροπής Προϋπολογισμών. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 15, παράγραφος 6, ε, α, νέο, καλύπτεται από το μπλοκ 3, άρα πάμε στο άρθρο 16 παράγραφος 1. Τροπολογία 45 της κυρίας Αρκίνη, Πέρ. κατά, αποχές, εγκρίνεται, να υπαλληθεύσουμε. Ναι, όχι, όχι. Ωραία. Τροπολογία 274 και 5 καταπίπτουν και πάμε στην παράγραφο 3 του άρθρου 16, 46 τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα παράγραφος 4, τροπολογία 276, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47 της εισηγήτριας υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά το 16, παράγραφος 4, τροπολογία 217, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 6, παράγραφος, άρθρο 16, παράγραφος 6, 48, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Άρθρο 18, παράγραφος 1, β, 279 της κυρία Ζούμπερ, υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. Άρθρο 18. Α, όχι, να επαληθεύσουμε. Την 279. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Νίκος υπέρ, 20 κατά. Δεν υιοθετείτε. Λυπούμε, κυρία Σούμπερ. Και τώρα ψηφίζουμε το 16 των γυναικών υπέρ. Κατά αποχές δεν ξέρω. Ψηφίζουμε την παράγραφο 16 της Επιτροπής Γυναικών. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 20 υπέρ, 21 κατά. Δεν εγκρίνεται. Και περνάμε στην 280 της κυρίας Κορνέλισεν. Ποιος είναι υπέρ. 280 τροπολογία της κυρίας Κονέλης είναι η είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 280 δεν εγκρίνεται. Άρα το Β δεν τροποποιείται. Άρα το 18 παράγραφο 2. 281. Τόμας Μαν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 18. Μετά την παράγραφο 3. 17 γυναικών υπέρ κατά αποχές. Η 17 εγκρίνεται άρθρο 19 και τον τίτλο τροπολογία 50 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18.1 πρόκειται η συμβαστική ΑΕ, 5 πολιτικές ομάδες ε, υποστηρίζουν υπέρ κατά το ΑΕ, συμβαστική τροπολογία εγκρίθηκε. 19-2 Πρόκειται για την 7. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 21α. Προϋπολογισμών. Υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε. Τέλος. 33 υπέρ 8 κατά. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το άρθρο 20, παράγραφος 1, σημείο Β, την 51 προϋπολογισμών υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20 άρθρο παράγραφος 2, 8 του ελέγχου προπολογισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 20 μετά την παράγραφο 2 πρόκειται για την 26 ίντα και 40 περιφερειών. Ταυτόσημες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 21 παράγραφος 1 σημείο α παράγραφος 20 γυναικών υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. Λοιπόν, κάτι δεν έκανα καλά. Θα πρέπει να επιστρέψουμε και να ψηφίσουμε κάποιες τροπολογίες που ήταν συμβατές. Το άρθρο 20, παράγραφος 1β, Παράγραφος 19 της Επιτροπής Γυναικών. Κατά εισηγήτρια ποιος είναι υπέρ. 19-19 των γυναικών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η 19 των γυναικών. Κατόπιν στην επόμενη παράγραφο η 284 της κυρίας Μπάουερ που είναι συμβατή με το 8 υπέρ της 284 κατά αποχές εγκρίνεται η 284. Να ελέγξουμε την 284 της κυρίας Μπάουερ. Πέρα στις πληροφορίες. 18 υπέρ, 23 κατά, 0 αποχές, κάτι άλλαξε. Και τώρα περνάμε στην 21, παράγραφος 1, γυναικών 21 υπέρ, κατά, αποχές, υπέρ, υπέρ της 21, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 9 ελέγχου προπολογισμού υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 παράγραφος 3 285 της κυρίας Σούμπερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 παράγραφος 4 υπό παράγραφος 1 πρόκειται για την 10 του ελέγχου προπολογισμού υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 της ίδιας επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 22 παράγραφος 4. 286 της κυρίας Σούμπερ. Υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. 286. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 286. Άρθρο 23. καλύφθηκε. 24, 2, 12 του ελέγχου προπολισμού υπέρ. Όχι, όχι, όχι, καλύφθηκε και αυτό, συγγνώμη, από τον μπλοκ 3. Περνάμε λοιπόν στην παράγραφο 1 των προπολογισμών υπέρ. Προϋπολογισμών 1, παράγραφος 1, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Και πάλι με δεύτερη παράγραφος που έχει προτείνει η Επιτροπή Προπολογισμών, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Κατόπιν, η συμβαστική α, πέντε πολιτικές ομάδες, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Μετά το 2, τροπολογία 60 της κυρίας Μπιζότο σε δύο τμήματα. Η ομάδα των σοσιαλιστών προτείνει να σταματήσει η φράση μετά αγορά εργασίας, labor market. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος της 60, υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. Άρα μπορούμε να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα μόνο του, Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ε, Για την αιτιολογική σκέψη 3, τροπολογία 65 της κυρίας Κορνέλησεν, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 3 της Επιτροπής Προϋπολογισμών, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δύο, της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την ιδεολογική σκέψη 3, 66, Νταρντέν, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συγγνώμη, λέει η πρόεδρο, θα πρέπει να ψηφίσουμε και την παράγραφο 4 τη Επιτροπή Προπολογισμών. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Για την αιτιολογική σκέψη 4 ψηφίζουμε τη δεύτερη συμβαστική πρόταση 6 ομάδων. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά τη αιτιολογική σκέψη 4 Τροπολογία 71. Τζούμπερ. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα μέχρι χιλιάδες εργασίες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Για το υπόλοιπο τμήμα το δεύτερο, το υπόλοιπο κείμενο υπέρ, κατά. Θα πραγματοποιήσουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 71 της κυρίας Ζουμπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται με 17 ψήφους υπέρ και 24 κατά. Το δεύτερο τμήμα λοιπόν της τροπολογίας 71 απορρίπτεται. Μετά το 4 έχουμε την συμβαστική ε, ε, J. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά τη αιτιολογική σκέψη 4 έχουμε την παράγραφο 2 τη επιτροπή Γυναικών υπέρ. Κατά αποχέ. εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 5, τροπολογία α, α, καλύπτεται. Μετά την αιτιολογική σκέψη 6 τώρα έχουμε την τροπολογία 7 της Επιτροπής Προπολογισμών. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές Εγκρίνεται η παράγραφος 7 της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Για την ιτολογική σκέψη 7 ψηφίζουμε την τρίτη συμβαστική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται η συμβαστική σε. Μετά την αιτιολογική σκέψη 7 έχουμε την παράγραφο 4 Επιτροπής Γυναικών ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικό έλεγχο για την παράγραφο 4 τη Επιτροπή Γυναικών. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Ισοπαλία 20 περί 20 κατά και μία αποχή. Άρα απορρίπτεται η παράγραφος 4 της Επιτροπής Γυναικών. Καλώς έγινε ο έλεγχος. Περνάμε τώρα στη συμβιβαστική δέλτα για την αιτιολογική σκέψη 9 από 6 ομάδες. Ποιος είναι υπέρ. Α, δεν ψηφίζουμε λέει η πρόεδρος γιατί εντάσσεται σε ένα μπλοκ. Τώρα για την αιτιολογική σκέψη 10 ψηφίζουμε τη συμβαστική ε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 11 Συμβαστική F από 6 ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 J, J από 6 ομάδες ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική H από 6 ομάδες ποιος είναι υπέρ κατά αποχές για την αιτιολογική σκέψη 13 εγκρίνεται. Μετά τη 13 έχουμε την τροπολογία 110 που καλύπτεται. Οπότε ψηφίσουμε για την αιτιολογική σκέψη 14 την συμβαστική I από πέντε πολιτικές ομάδες. Δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε γιατί καλύπτεται από τον μπλοκ 4 που ήδη ψηφίσαμε. Οπότε ψηφίζουμε την τροπολογία 115 για την ιδεολογική σκέψη 15. Είναι τροπολογία Bauer. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 115. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορία. Ψήφισαν 13 υπέρ, 25 κατά και 3 αποχές. Απορρίπτεται λοιπόν η τροπολογία 115. Σας ευχαριστώ για την επαγρύπνηση και την εγρήγορσή σας. Ψηφίζουμε τις τροπολογίες 12 Χάρκιν και 116 Κορνέλισεν που είναι πανομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνονται. Αιτιολογική σκέψη 16. Οι τροπολογίε αυτές εντάσσονται στο μπλοκ 3, οπότε δεν χρειάζεται να τι ψηφίσουμε. Μετά την αιτιολογική σκέψη 16, παράγραφος 18 της Επιτροπής Προϋπολογισμών, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Για την αιτιολογική σκέψη 18, παράγραφος 19 της Επιτροπής Προϋπολογισμών, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 120, Κάμπρνοχ, συμβατή. Ψηφίζουμε λοιπόν Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Για την αιτιολογική σκέψη 19, παράγραφος 20 Επιτροπής Προϋπολογισμού, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά το 19, τροπολογία 121, κορνέλησεν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 19 και πάλι, αιτιολογική σκέψη 19 μάλλον, Τροπολογία 122 καταπίπτει, οπότε φτάνουμε στην αιτιολογική σκέψη 21 και την παράγραφο 21 της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ολοκληρώσαμε την ψηφοφορία των τροπολογιών μας και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, παρακαλώ, το σύνολο της έκθεσης κυρίας Χάρκιν. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η έκθεση με 35 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 3 αποχές. Ψηφίζουμε τώρα το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 35 ψήφισαν υπέρ, 2 κατά και 3 αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Χάρκιν. Δεν είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα με την Επιτροπή Γεωργίας. Ο κύριος Όρη, διαδικαστικό. Ε, ε, mert más mutattam és más nyomtam véletlenül, tehát a, gomb negatívat mutatott, de én pozitívat, tehát plusz szavaztam. Εγώ ψήφισα ναι, αλλά βλέπω ότι έχει καταμετρηθεί σαν όχι. Ήθελα να το πω εκείνη την ώρα, αλλά δεν πρόλαβα. Βάλτε σας παρακαλώ ένα συν στο όνομά μου και όχι μείον. Προσπάθησα να το διορθώσω, αλλά η μηχανή δεν υπάκουσε. Euh, Μα δεν σας ακούει και η μηχανή, τι να σας πω. Αυτό ήταν στο σχέδιο νομοθετικού περιεχομένου, στο σχέδιο έκθεσης. Ωραία, άρα ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία για την εισηγήτρια, την κυρία Αρκίνη. Σας παρακαλώ πολύ. Ένα λεπτό ακόμη. Μετά τη ψηφοφορία αυτή μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο προκειμένου να υλοποιηθεί συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με, βάση το άρθρο 70 παράγραφο 20, παράρτημα 21 του κανονισμού μας και να σας επισημάνω ότι δεν θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις με την Κυπριακή Προεδρία γιατί η Κυπριακή Προεδρία δεν επιθυμεί να οργανώσει τριμέρις διαλόγους μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Οπότε προτείνω να περιμένουμε τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα στις 28 ε, Νοεμβρίου με θέμα το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και μάλιστα και θα κριθεί και το μέλλον του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και τότε θα αποφασίσουμε αν θέλουμε όντως να εγκαινιάσουμε να με το Συμβούλιο για συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση ή μήπως προτιμάμε να παραπέμψουμε την ψηφοφόρια στην Ολομέλεια. Ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα, τώρα ως προς το χρονοδιάγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έκανα λάθος, ε, θα είναι 20 με 23 Νοεμβρίου, Οπότε στη δική μας συνεδρία στι 18 και 19 Νοεμβρίου θα λάβουμε απόφαση για το τι θα γίνει ανάλογα και με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αν δεν υπάρχουν διάφορα, ολοκληρώσαμε ραντεβού στις 13 Νοεμβρίου. Και θα έχουμε μία κοινή συνεδρίαση με τον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας, ε, κοινή συνεδρίαση με την Οικονομική Επιτροπή και φυσικά περιμένω να είστε όλοι παρόντες εκεί. Καλώς βράδυ.